Κύριε Πρόεδρε Μπουχάρη, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να καλωσορίσω εκ βάθου καρδία τον πρόεδρο τη Νιγηρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Μπουχάρη. Πριν από ένα χρόνο σχεδόν εξελέγεται ως πρόεδρος της Νιγηρίας μετά από μια ειρηνική και δημοκρατική διαδικασία και έχετε προχωρήσει σε μια πάρα πολύ πλήρη και φιλόδοξη ατζέντα μεταρρυθμίσεων για να αντιμετωπιστούν τα θέματα της λειτουργία του κράτους και διαφθοράς στην Ιγυρία και να, αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπιστεί και η μαστίγα της τρομοκρατίας. Μετά από τις φρικτές ενέργειες και ομότητες του Μπόκο Χαράμ που είναι στη συνείδηση όλων μας. Μετά από τη σειρά αυτή επιθέσεων και της τελευταίας εβδομάδας που με τους τωρινούς με τα τωρινά στοιχεία έχουν χάσει τη ζωή τους 85 άτομα εμείς θέλουμε να τονίσουμε την αλληλεγγύη μας προς τον λαό της Νιγηρίας Έχω διαβεβαιώσει τον πρώτο Μπουχάρη ότι και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε μαζί του στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Και φυσικά υποστηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα του και είμαστε έτοιμοι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσουμε τον πρόεδρο Μπουχάρη και την Ιγυρία για να υπάρξει και οικονομική ανάπτυξη και επενδύσεις στην χώρα αυτή. Θα εξονόματος λοιπόν των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σας ε, καλωσορίζω κύριε Μπουχάρη, κύριε Πρόεδρε και σας ζητώ να λάβετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Σούλτς, κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί κύριοι βουλευτές, διακεκριμένοι κύριοι και κυρίες. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Μάρτιν Σούλτς, για την πρόσκληση που μου απίφθινε να λάβω το λόγο ενώπιον της ε, Ολομέλειας του νομοθετικού αυτού σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί για μένα μια μεγάλη τιμή και με ταπεινοφροσύνη θα χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία να λάβω το λόγο ενώπιον σας. Θέλω επίσης να τονίσω προς τους ηγέτες της Ευρώπης, προς τους κοινοβουλευτικούς, προς όλους τους ανθρώπους της Ευρώπης, θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα καλής θέλησης από τους συμπατριώτες μου. Ο λαός της Νιγηρίας αναγνωρίζει και εκτιμά ιδιαίτερα τις υλικέ και χρηματικές θυσίες τις οποίες έχει υποστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα φιλικά έθνη της Ευρώπης για να μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι εκλογές και η προώθηση και εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών στην Ιγυρία. Όπως είχε πράξει και στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει την ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή στην Ιγυρία για να μπορέσουν να λάβουν χώρα με ομαλό τρόπο οι γενικές εκλογές στην Ιγυρία και το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών έγινε αποδεκτό από όλη τη διεθνή κοινότητα με ικανοποίηση. Η Ιγυρία καταγράφει τη σημαντική συμβολή που έχει κάνει η Ευρώπη προς την επίτευξη ικανοποιητικών, ελευθέρων και δίκαιων εκλογών στην χώρα μας και αμερόληπτων εκλογών. Σήμερα μπορώ να τονίσω στο ενώπιον του σώματός σας ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις αρχίζουν να καρποφορούν. Είμαι ένας από τα αποτελέσματα, ένας από αυτούς οι οποίοι ε, μπόρεσαν να προκύψουν από αυτήν τη διαδικασία δημοκρατικοποίησης στην Ιγερία. Το τωρινό καθεστώς λοιπόν είναι και το αποτέλεσμα δημοκρατικών επιλογών που έγιναν με απόλυτη επίγνωση από το λαό της Νιγηρίας μέσω των, καλ, των καλπών και των εκλογών. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε και κύριοι, η δημοκρατία έχει έλθει και θα παραμείνει στην Νιγηρία. Πολύ πιο νωρί από ό,τι πολλοί από εμά είχαμε φανταστεί. Η Νιγηρία θα είναι μία από τις πιο σταθερές, ισχυρές και εύρωστες δημοκρατίες στην Αφρική. Μπορούν να εξακολουθούν να υπάρχουν αντιπαραθέσεις και εντάσεις, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν και να παραμείνουν μέσα στο πλαίσιο των μηχανισμών ασφαλείας μιας εκλογική δημοκρατία που βασίζεται σε εκλογέ. Τα γεγονότα που οδήγησαν στι γενικέ εκλογέ τη Νιγηρία στι αρχέ του 2015 είχαν καταρχήν δείξει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στη χώρα μου υπήρχε ένα κλίμα οργής, υπήρχαν αντεγκλήσεις και αντιπαραθέσεις, υπήρχαν εχθρικές ενέργειες, απειλές, βία που χρησιμοποιήθηκε εναντίον των εκλογέων με στόχο να τους υποχρεώσει να ψηφίσουν για το τότε καθεστώς, το status quo. Όλα αυτά ήταν εξελίξεις πάρα πολύ αρνητικές που έθεταν αναμφιβόλο τη σταθερότητα της Νιγηρίας. Τα δραματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην, στο Εθνικό Κέντρο Συγκεντρωτικής Καταμέτρησης ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν πραγματικά τρομακτική και ήταν το αποτέλεσμα ενεργειών ε, πρακτόρων του καθεστώτος, του τότε καθεστώτος, μέσα στα πλαίσια της απόγνωσής τους για να μπορέσουν να διατηρήσουν την, τον θανάσιμο εναγκαλισμό τους στους εθνικούς πόρους για λόγους καθαρά εγωιστικούς η υπομονή και η οριμότητα με την οποία οι αξιωματούχοι της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής υπό τον καθηγητή Αταχύρου Χίγκα μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό, διέσωσαν τη δημοκρατία και δικαίωσαν την Μεγάλη Ευρωπαϊκή Συμβολή θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό για το γεγονός ότι η Νιγηρία μπόρεσε να βγει άμομη από αυτή τη δραματική κατάσταση. Όπως τόνισε και σε άλλους χώρου, η δράση του προηγουμένου Προέδρου της Νιγηρίας, του Γκουτλακ Έμπελε Γιώναθαν, είναι επίσης αξιέπαινη. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της Νιγηρίας ένας εξερχόμενος πρόεδρος και υποψήφιος για την Προεδρία παραδέχτηκε την εκλογική ήττα του παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί οι οποίοι του ζητούσαν να παραμείνουν στην εξουσία. Πολλοί από τους πράκτορες και από αυτούς που ωφελήθηκαν από την προηγούμενη κατάσταση. Αγαπητοί κύριοι κοινοβουλευτικοί, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για την ειδική σχέση που υπάρχει μεταξύ της Νιγηρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος εταίρος ανάπτυξης της Νιγηρίας και ένας πυλώνας υποστήριξης για την εδραίωση της δημοκρατίας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας. Κύριε Πρόεδρε, εμείς προερχόμενοι από την Αφρική εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα δικά σας προβλήματα είναι κυρίως η διαχείριση της ευμάρειας και του ανταγωνισμού. Αντίθετα, τα δικά μας προβλήματα είναι η ένδια, η ασθένεια, η τεχνολογική υστέρηση. Δεν είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς τα προβλήματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν για μας. Έχουμε εσωτερικές αντιπαραθέσεις, κύματα προσφύγων, ανθρώπους που προσπαθούν να διαφύγουν με βάρκες, την αλαθρεμπορία ε, ανθρώπων και ναρκωτικών και όλα αυτά. Το χάος αυτό δεν είναι κάτι που θα το ζήλευε οποιοδήποτε από τους γείτονές μας. Γι' αυτό είναι προ το κοινό μα συμφέρον να συνεργαστούμε και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στην Αφρικανική Ήπειρο. Χαίρομαι κύριε Πρόεδρε για το γεγονό ότι υπάρχει ήδη ο ετήσιο πολιτικό διάλογο μεταξύ Νιγηρία και Ευρωπαϊκή Ένωση, και μέσω αυτού του διαλόγου έχουμε συνεχίσει να ενισχύουμε τη συνεργασία μα, η οποία βασίζεται σε κοινέ αξίε και κοινά συμφέροντα ιδίω σε ό,τι αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη δημοκρατία και την ευκυβερνησία. Μέσω αυτού του φόρουμ έχουμε επιτύχει τη συνέχιση σε τακτική βάση των κοινών μας προσπαθειών για να έχουμε κοινέ κατευθύνσεις σε σημαντικά περιφερειακά, υπηρετικά και παγκόσμια θέματα με στόχο την επίτευξη κοινών θέσεων. Είμαστε προσιλωμένοι στην εντατικοποίηση του πολιτικού αυτού διαλόγου και της συνεργασίας στα πλαίσια <clears throat> της κοινή πορεία της Νιγηρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο πλευρές πιστεύουν στην ειρήνη και την ασφάλεια, στο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την σωστή διακυβέρνηση, την ισότητα, την ανεκτικότητα, γιατί όλοι αυτοί είναι οι σωστοί δρόμοι για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ευμαρείς και ισχυρές κοινωνίες. Επιπλέον, στα πλαίσια αυτής της ίδιας σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νιγηρίας, θα ήθελα να αναγνωρίσω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει με πολύ αυστηρό τρόπο καταδικάσει τις ενέργειες εξτρεμιστικών ομάδων μεταξύ των οποίων της Μπόκο Χαράμ στην Νιγηρία και στην, ε, στο σύνολο της ε, κοινότητας των δυτικοαφρικανικών κρατών, της ECOWAS. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταγράψει και έχει επενέσει την ανάπτυξη στην Ιγυρία μιας εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής και της τροποποιήσεις στον εθνικό αντιτρομοκρατικό νόμο ως ε, δείγμα της ε, δέσμευση της κυβέρνησή μα να βρούμε μια μόνιμη λύση στι απειλές του Μπόκο Χαράμ. Η Νιγηρία χαίρεται για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίω στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης, της δημιουργίας ικανοτήτων για τις δυνάμει ασφαλεία και επίση την παροχή αρρωγής για ανάπτυξη. Από τη δική μας πλευρά, εμείς έχουμε τροποποιήσει <clears throat> τους κανόνες εμπλοκής σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και έχουμε αποδώσει πολύ μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της, των δρασεών μας στην αντιμετώπιση των εχμαλωτιστέντων τρομοκρατών, των πολιτών που έχουν εμπλακεί στις αντιπαραθέσεις αυτές και γενικά στην διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών μας. Ο στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την ελάχιστη δυνατή βία για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Εν ώψη όλων αυτών, θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τα μεμονωμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δώσει βοήθεια προς τις νιγηριανές στρατιωτικές δυνάμεις ώστε να αντιμετωπίσουν τα τρομοκρατικά στοιχεία του Βοκοχαράν. Πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποσχεθεί να υποστηρίξουν τις προσπάθειές μας προς την ε, διάσωση των απαχθέντων κοριτσιών της σχολής Τσίμποκ. Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει ότι σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε τους γονείς αυτών των κοριτσιών τους διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή μας δεν θα αφιστεί προσπαθειών μέχρι ότου διασωθούν ζωντανές όλες αυτές οι κοπέλες και επανέλθουν στις οικογένειές τους παραμένω απόλυτα δεσμευμένος για την επίτευξη αυτού του στόχου. Μετά από την ανάληψη εξουσίας τον Μάιο του προηγούμενου έτους έχουμε αναδιοργανώσει τις ένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας και τις έχουμε αναδιατάξει ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον, την τρομοκρατία του Μπόκο Χαράμ όλες οι τοπικές κυβερνητικές περιοχές που στο παρελθόν ήταν υπό τον έλεγχο του Μπόκο Χαράμ, στο Ανταμάουα, στο Μπόρνο και στο Γιόμπε, στο Ανατολικό τμήμα της Νιγηρίας, έχουν ανακτηθεί από τις κυβερνητικές δυνάμεις τα οι εσωτερικά εκτοπισμένοι της Νιγηρίας επανέρχονται σιγά σιγά στις αιστείες τους. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας είναι προσιλωμένη στην ανοικοδόμηση σχολείων, νοσοκομείων και άλλων ζωτικών στοιχείων υποδομής που έχουν καταστραφεί από τους αποχωρούντες τρομοκράτες. Αυτή τη στιγμή η δράση του Μπόκο Χαράμ έχει περισταλεί μονάχα στο δάσος του Σαμπίσα και η ικανότητά τους να ξεκινήσουν επιθέσεις μεγάλης κλίμακος έχει μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά. Το Μπόκο Χαράμ τώρα μονάχα αντιμετωπίζει και επιτίθεται σε εύκολους στόχους όπως είναι οι αγορές, τα ζαμιά και οι εκκλησίες χρησιμοποιώντας αθώα και άτυχα ε, ανήλικα παιδιά για να για να πυροδοτήσουν τοπικά κατασκευασμένα αυτοσχέδια κριτικά μηχανίσματα. Επίσης πρέπει να εκφράσω την σοβαρή ανησυχία μας για την επικίνδυνη κατάσταση στην Νότιο Λιβύη που γίνεται μια στρατηγική ορολογική βόμβα για την Αφρική και την Ευρώπη. Οι ακυβέρνητες περιοχές ε, της Νότιας Λιβύης ε, έχουν γίνει ένα αποδοτικό παζάρι όπλων που απειλεί την ασφάλεια της περιοχής του Σαχέλ και της Σαχάρα, αλλά ολόκληρη την Δυτική Αφρική και πέραν αυτή. Κατά συνέπεια πρέπει να, εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για να βρεθούν μόνιμες λύσεις στην κρίση της Λιβύης. Κύριε Πρόεδρε, η Νιγηρία είναι ένα φιλιρνικό έθνος και έχει παίξει ένα κρίσιμο ρόλο στην διαχείριση και επίλυση σειράξεων εντός και εκτός της Αφρικής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Κυρίε και κύριοι, η διατήρηση και η οικοδόμηση της ειρήνης αποτέλεσαν τμήμα της εξωτερικής πολιτικής της Νιγηρίας από την ανεξαρτησία της. Οι δυνάμεις της χώρας μετέσχουν σχεδόν σε όλες τις ε, αποστολές ειρήνης σε υποεθνικό, υποπεριφερειακό και περιφερειακό επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών και παρά τις προκλήσεις στην ασφάλεια που αντιμετωπίζουμε τώρα, έχουμε συμβάλει, είμαστε μεταξύ των 10 χωρών που έχουν συμβάλει περισσότερο στις ειρηνευτικέ διαδικασίες του ΙΕ ανά τον κόσμο, με, τεράστιο, με τεράστια δέσμευση, τόσο οικονομική όσο και σε ανθρώπινους πόρου. Η πρώτη εμφάνιση τη Νιγηρία σε ειρηνευτική διαδικασία ήταν στο Κονγκό, ω μέλο ε, τη ε, δύναμη των Ηνωμένων 20.000 ατόμων της ΟΝΟΚ τον Ιούλιο του 1960. Είχα την τιμή να είμαι και μέλος στο, στην Ιγυριανή δύναμη του 1963. Αυτό ήταν τρεις μήνες μόνο μετά την, πριν την ανεξαρτησία της Νιγηρίας. Μετήχαμε επίσης στις ε, επιχειρήσεις του ΙΕ στο Κονγκό για 3,5 χρόνο, χρόνια. Συμβάλαμε στο Κονγκό ως η τρίτη μεγαλύτερη εθνική ομάδα μετά του Ινδού και τις Οθίωπε. Έκτοτε η Νιγηρία παραμένει και διατηρεί μία παρουσία στις παγκόσμιες ειρηνευτικέ προσπάθειες και μάλιστα έχει μετάσχει στην διατήρηση του νόμου και της τάξης μετά από μία ανταρσία στην Ταγκανίκα το 1964, το 1979 και το 1982 στρατιώτες του 21ου τάγματος πεζικού της Νιγηρίας και του 200ου δευτέρου συντάγματος αναγνώρισης είχαν στάλει στο Τσάντ ως ειρηνευτική δύναμη για την παρακολούθηση της εκεχηρίας παρέχοντας εμπιστοσύνη στην συνεχιζόμενη ειρηνευτική διαδικασία. Επιπλέον συνέβαλε με την, ως μεγαλύτερη, μεγαλύτερο τμήμα στις ε, δυνάμεις της οικονομικής κοινότητας της Δυτικής Αφρικής στην παρουσία της στην στη Σιέρα Λεόνε. Η οικονομική κοινότητα των χωρών της Δυτικής Αφρικής με την ομάδα παρακολούθησης αποκατέστησε την τάξη στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας και επέστρεψε τον διοχθέντα πρόεδρο Τέιαν Κάμπα στα, στα καθήκοντά του στις 10 Μαρτίου του 1998. Υπό την εντολή της Αφρικανικής Ένωσης η Νιγηρία ξεκίνησε μια ειρηνευτική αποστολή στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε όπου κατόρθωσε να πείσει αντάρτες στρατιώτες να υπακούν στις συνταγματικές αρχές. Επιπλέον η Νιγηρία απέστειλε προσωπικό στη Ρουάντα και στην περιοχή του Νταρφούρ του Σουδάν για τη διατήρηση της ειρήνης στις δύο αυτές χώρες. Πρόεδρε, η Νιγηρία επιπλέον έχει, στάλει, έχει στείλει δυνάμεις στις ακόλουθες αφρικανικές χώρες. Στην Αγγόλα, στην ε, αποστολή επαλήθευσης των Ηνωμένων, Εθνών στην ε, Αγγόλα, στην Αμίμπια, στην ομάδα ε, επικουρίας της χώρας, στη Μοζαμβίκη, στη Δυτική Σαχώρα, στη Σαχάρα, στην αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα, στη Σομαλία, στην, στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών στην Σομαλία και στην Λοίδα του Αούζου, στην ομάδα παρατηρητών του ΟΗΕ για το Αούζου. Κυρίε και κύριοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το θέμα της μετανάστευσης από την Αφρική στην Ευρώπη. Η Νιγηρία αναγνωρίζει και συμμερίζεται τις ανησυχίες που έχει εκφράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με μη ζωή μεταναστών από την Αφρική μέσω της Μεσογείου και με τις συνεπαγόμενες απώλειες ζωών. Προς τούτο η Νιγηρία θα συνεργαστεί με την Αφρικανική Ένωση για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης στην Ευρώπη. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τον παράγοντα παρότρινσης της μετανάστευσης, ιδίως από την Νιγηρία και ως χώρα τράνζιτ ε, ε, και ως χώρα αποστολής. Στον προϋπολογισμό της χώρας φέτος η κυβέρνηση προβλέπει 500.000 θέσεις εργασίας μόνο στον τομέα της, ε, των εκπαιδευτικών. Συνεργαζόμαστε επίσης με τις πολιτείες και την τοπική αυτοδιοίκηση για να ενισχύσουμε τα κέντρα κτήσης δεξιοτήτων, ούτως ώστε να εκπαιδεύσουμε τους νέους σε, διάφορα, σε διάφορες δεξιότητες και προσόντα για να μπορούν να βρουν θέση για να μπορούν να βρουν δουλειά και να γίνουν με τη σειρά τους εργοδότες. Επίσης καταβάλουμε προσπάθειες για να διαφοροποιήσουμε την οικονομία, παροτρύνοντας στην, δίνοντας έμφαση στην γεωργία, στα στερεά ορυκτά και την εκμετάλλευσή τους για να δημιουργήσουμε πλούτο και θέση εργασίας. Η Νιγηρία καλωσορίζει την έκβαση της Συνόδου Κορυφής Ένωσης Αφρικής στη Βαλέτα για την ε, μετανάστευση, μεταξύ των οποίων και το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης ε, ύψους ενός δισεκατομμυρίου 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των βασικών αιτιών μετανάστευσης από την Αφρική στην Ευρώπη. Η Νιγηρία θα συνεργαστεί με τις χώρες του Σαχέλ και της Κεντρικής Αφρικής υποβάλλοντας στο Συμβούλιο του Ταμείου αυτού έκτακτης ανάγκης τα έργα που έχουμε στοχοθετήσει για τη χρηματοδότηση. Η κοινή ημερήσια διάταξη για τη μετανάστευση και την κινητικότητα που υπέγραψε η Νιγηρία στις 12 Μαρτίου 2015 ήταν και μάλιστα ήταν η πρώτη χώρα που είχε υπογράψει αυτή τη συμφωνία από πλευράς ε, υποσαχάριας Αφρικής. Τούτο αποτελεί απόδειξη του θετικού πνεύματος συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της μετανάστευσης και της ανάπτυξης. Υπό το φως αυτής της επίγνωσης είναι που θέλω να προτείνω την αμοιβαία άρση θεωρήσεων για τους ε, κατόχους διπλωματικών και επισήμων διαμαρτυρίων της Νιγηρίας που προέρχονται σε επίσημες συναντήσεις και διασκέψεις στην Ευρώπη. Τώρα για το θέμα των συμφωνιών εταιρική συνεργασίας. Η Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και της Ομάδας των Χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού και που έχουν συλλογικά υποστηριχθεί από την οικονομική κοινότητα των χωρών της Δυτικής Αφρικής δεν έχει ακόμα υπογραφεί από την Ιγυρία και κάποιους άλλους. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την Συμφωνία Οικονομικής ε, Συνεργασίας η Νιγηρία έθεσε μια σειρά σημαντικών τεχνικών ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεδομένης ε, της ε, ανισορροπίας μεταξύ των δύο περιφερειών Ευρώπη και σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και την εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα, η Ένωση Κατασκευαστών της Νιγηρίας και οι συνδεδεμένες ε, εργοδο... Ε, ε, οργανώσεις εργαζομένων έδεσαν ανησυχίες για τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν αυτές οι συμφωνίες στο πρόγραμμα εκβιομηχάνησης της Νιγηρίας. Η Νιγηρία αγωνίζεται για να αντιμετωπίσει από πλευρά τα δύο αυτά ζητήματα. Ζητώ λοιπόν από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν και αυτοί από πλευρά τους τις ανησυχίες μας επιτρέποντας η Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας να είναι αμοιβαία επωφελής και να συμβάλλει στην ευημερία των λαών μας στο πλαίσιο των κοινών αξιών και συμφερόντων για να προωθήσουμε εγκάρδιες διμερές εμπορικές σχέσεις. Κλοπή πετρελαίου και παράνομη αποθήκευση καυσίμων. Η Νιγηρία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλοπής πετρελαίου και της παράνομης αποθήκευσης ε, καυσίμων στο δέλτα του Νιγήρα, καθώς και την ανάκτηση των παρανόμως κτηθέντων πόρων. Είναι σκόπιμο λοιπόν να τεθούν τα θέματα αυτά ενώπιόν σας, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές. Η Νιγηρία στο θέμα αυτό ζητά την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξη των προσπαθειών που έχουν στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Η προσπάθειά μας να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια, να περιορίσουμε την διαφθορά και να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα θα οδηγήσει προφανώς στη βελτίωση της κοινωνικής σταθερότητας στην Ιγυρία, αλλά θα ξανανοίξει τις πόρτες για πλήρες οικονομικές σχέσεις με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο αυτοί που θέλουν να επενδύσουν στις χώρες μας έχουν τεράστιες ευκαιρίες και προτιθέμεθα να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των ατόμων και των επενδύσεων που έρχονται στην Νιγηρία. Κύριε Πρόεδρε, ο κόσμος πρόσφατα, ολόκληρος ο κόσμος πρόσφατα συναντήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας στη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος, την COP21. Η θετική αντιμετώπιση του θέματος οδήγησε σε αμοιβαία αποδεκτές αποφάσεις. Οι ηγέτες όλου του κόσμου υιοθέτησαν μια κοινή πλατφόρμα για να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, ιδίως στις λιγότερο ε, στις πιο μειονεκτούσες χώρες ανά τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της πολύ σημαντικής αυτής παγκόσμιας εκδήλωσης δήλωσα την θέση της χώρας μου ως προς την αλλαγή του κλίματος. Επαναλαμβάνω εδώ ότι ενέχει σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και ανάπτυξη της Νιγηρίας. Η Νιγηρία παρακολουθεί αβοήθητη την αποξήρανση της λίμνης Τσάδ. Αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στον κόσμο που ζει εκεί και που για γενιές στηριζόταν για την διαβίωσή τους τους πόρους της λίμνης. Πόρους που σιγά σιγά και που πολύ γρήγορα εξαφανίζονται διώχνοντας ε, από τις θέσεις εργασία μια σειρά κοινοτήτων. Πρόεδρε, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι παρόχθιες χώρες της λίμνης Τσάντα αντιμετωπίζουν όλες τις επιπτώσεις αλλαγής του κλίματος. Συλλογικά είμαστε υπό την υποχρεώση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινέ αλλαγέ. Οι συλλογικές μας προσπάθειες μπορεί να μην είναι αρκετές, καθώς είμαστε περιορισμένοι από την έλλειψη κονδυλίων, τεχνολογίας και ανθρώπινο δυναμικού για να ξεκινήσουμε και να υιοθετήσουμε τις σωστές λύσεις. Ζητούμε για το λόγο αυτό να υπάρξει δράση σε παγκόσμιο επίπεδο και γρήγορα για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών που θα συμβάλλουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την λίμνη του Τσάντ. Σε μια προσπάθεια να βρεθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα αυτό, η Νιγηρία συνέβαλε με 5 εκατομμύρια δολάρια ΙΠΑ που χρησιμοποιήθηκαν ήδη για την διαξαγωγή μιας ολιστικής μελέτης για τη μεταφορά νερού από την λεκάνη του Κόγκο στην λίμνη Τσάντ. Η μελέτη έδειξε ότι το έργο αυτό θα απαιτήσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια για να ολοκληρωθεί. Θέλω να αναφέρω ότι η μελέτη αυτή ανέφερε ότι το προτινόμενο έργο για τη λίμνη Τσάντ θα μπορέσει να αποπληρώσει την τεράστια αυτή επένδυση αν ε, χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, καλώ το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που έχει για να βοηθήσει στην ε, ενίσχυση της υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου αυτού. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω εκ νέου να εκφράσω με κάθε ταπεινότητα την βαθιά εκτίμησή μου προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τα μέλη του, την ευρωπαϊκή Υγεσία και τον λαό της Υπήρου αυτής για την τιμή που μου έκαναν προσωπικά και σε μένα αλλά και διεμού στον λαό της Νιγηρίας να απευθυνθώ στην Ολομέλεια μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες δημοκρατιών του κόσμου. Σας ευχαριστώ για αυτή τη σπάνια τιμή. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε Μπουχάρη για την ομιλία σας. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για, την, για τα χειροκροτήματα και την υποστήριξή τους που αποτελεί υποστήριξη στο δύσκολο έργο του Πρόεδρου Μπουχάρη στη χώρα του και πάλι θα ήθελα εξ ονόματος όλων των συναδέλφων να σας ευχαριστήσω κύριε Μπουχάρη για τον μεγάλο αγώνα της ε, χώρας σας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών. Σας ευχαριστώ και πάλι για την επίσκεψή σας.